Good morning, ladies and gentlemen. I would like to ask... Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να κάτσετε για να ξεκινήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Our Agora meeting, Agora Congress uh, for European citizens. It is our third meeting Πρόκειται για την τρίτη μας συνεδρίαση. Ξεκινήσαμε χάρη στον Ευρωβουλευτή κύριο Ονεστά. Μεγάλη, σπουδαία ιδέα είχε. Και η πρώτη συνεδρίαση ήταν γενικότερη, γενικότερο περιεχομένου για την ε, συνεδρίαση της για την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και γενικές παρατηρήσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, θα μιλήσουμε για κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλους μας τους πολίτες. Διότι η φτώχεια, η ανεργία είναι κάτι που δεν αποτελεί απλά πρόκληση, αλλά απειλή για κάθε μεμονωμένο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο αντιπροέδρους, την κυρία Ιζαμπέλ Ντουιγάν και τον ε, Ρίμπο Βότσεκ που κάθονται δεξιά μου και αριστερά μου, διότι διοργάνωσαν την αγορά και μας συγκέντρωσαν εδώ όλους για τρίτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε βέβαιοι ότι θα πρέπει αυτό να γίνεται κάθε χρόνο. Μία συνεδρίαση πολιτών στην ουσία. Διότι εσείς αντιπροσωπεύετε τους πολίτες μας. Με τον πιο άμεσο τρόπο. Εσείς ε, εκλέγετε τους εκπροσώπους σας στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά εσείς ως εκπρόσωποι, η ΜΚΟ, οι οργανώσεις των πολιτών, είστε οι άνθρωποι που βρίσκεστε πιο κοντά στους πολίτες μας. Πάντοτε, είτε ε, πρόκειται, για τις τοπικές κοινότητες, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσία σας λοιπόν εδώ είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον Επίτροπο Άντορ, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Από ό,τι κατάλαβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζει για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Και πέρυσι, το έτος της καταπολέμησης της στόχης και του κοινωνικού αποκλεισμού, μπορούμε να πούμε ότι στην ουσία η σημερινή συνεδρίαση συνοψίζει ολόκληρο το έτος που πέρασε και επίση μαζί μα βρίσκεται η κυρία Πρόεδρο Μπρεσόν. Καλώ ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο και ο Πρόεδρος Νίλσον. Που αντιπροσφέρει την, την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τόσο σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες και τόσο αντιπροσωπευτική των Ευρωπαίων πολιτών σε, στη σημερινή συνεδρίαση των Βρυξελών. Έχουμε ειδικέ ε, δυνατότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε 23 γλώσσες Μόνο ένα τέτοιο μέρος υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο, με 23 ομιλούμενες γλώσσες κάθε φορά που το επιθυμείτε. Έχουμε λοιπόν ε, διερμηνία. Μπορείτε να μιλήσετε στην μητρική σας γλώσσα. Και εγώ ο ίδιος μπορώ να μιλήσω στη γλώσσα μου, την μητρική, και θα αλλάξω τώρα και θα μιλήσω στη γλώσσα μου, τα πολωνικά. Drodzy goście, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Αγαπητοί εκπρόσωποι των οργανώσεων των πολιτών, πρόκειται για την τρίτη φορά που συναντώμαστε σήμερα εδώ. Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ε, μέσο διαλόγου ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες και το Ευρωκοινοβούλιο, ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τις οποίες οι εκπρόσωποι είναι εδώ μαζί μας. Το ίδιο το όνομα αγορά των πολιτών είναι μεγάλη σημασία διότι μας παραπέμπει στις ρίζες της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι δυνατή χωρίς την κοινωνία των πολιτών. Η αγορά είναι ένα μέρος όπου η κοινωνία πραγματικά μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματά της, να εκφράσει τις επικρίσεις της και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι τεράστια σημασία για όλους μας. Υπάρχουν γείτονε γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η κοινωνική αναταραχή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα όπως στην Τινησία τη Λευκορωσία. Πριν από 20 χρόνια την ίδια κατάσταση, η ίδια κατάσταση επικρατούσε στα Δυτικά Βαλκάνια και χάρη στην προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άνοιγμα δυνατότητας συμμετοχής σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων επικράτησε πλέον η ειρήνη στις ε, περιοχές αυτές. Εχθές είχα μια σημαντική επαφή με τον επικεφαλής του Σερβικού Κοινοβουλίου. Η Σερβία παίζει σήμερα πολύ σημαντικό ρόλο ρυθμιστή στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη Αυτό είναι το ευρωπαϊκό σχέδιο, το ευρωπαϊκό όραμα. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί έχει τεράστιες θετικές επιπτώσεις στην ζωή των γειτονικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής είχαμε δύο συναντήσεις της πρωτοβουλίας της αγοράς των πολιτών. Μιλήσαμε για προβλήματα όπως οι κλιματικές αλλαγές. Σήμερα μιλάμε για την κρίση και τις διάφορες μορφές, τα διάφορα πρόσωπα της φτώχειας. Η οικονομική κρίση επηρεάζει τις ζωές σε πολλών Ευρωπαίων πολιτών. Δεν γινόμαστε πιο πλούσιοι, γινόμαστε πιο φτωχοί και χάρη σε εσά μπορούμε να εξεύρουμε τους τρόπους για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Γιατί οι πολίτες μας έχουν κάθε δικαίωμα να αναζητήσουν τη βοήθειά μας. Οπότε θα πρέπει εμείς να βρούμε τους τρόπους για να αποφύγουμε τέτοιες κρίσεις στο μέλλον, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σήμερα, σήμερα και όχι αύριο. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη με τους συμπολίτες μας. Και χρησιμοποιώ τη λέξη αλληλεγγύη γιατί αυτό αποτελεί φόρο τιμή στην συμμετοχή μου στο Συνδικάτο Αλληλεγγύη την δεκαετία του 80. Δέκα εκατομμύρια Πολωνοί πολίτες ε, υπό το κομμουνιστικό καθεστώς ε, μπήκαν σε αυτό το συνδικάτο μέσα σε δύο εβδομάδες. Δεν ξέραμε πώς και τι, πού θα καταλήγαμε. φοβόμασταν ότι μπορεί και να επιβληθεί στρατιωτικό νόμο, αλλά είχαμε το θάρρο να συμμετέχουμε στην ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτό το κίνημα που ήθελε να υπερασπιστεί την περηφάνεια των ε, πολιτών μας. Επίσης αγωνιζόμασταν για την ελευθερία της χώρας μας και όλων των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να δρά κανεί ως πολίτης και γι' αυτό και δημιούργησα ένα ίδρυμα για τα θέματα της υπηκότητας και κάθε χρόνο διοργανώνουμε έναν διαγωνισμό που χορηγεί βραβεία για τις καλύτερες πρωτοβουλίες πολιτών. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι γιορτάζουμε 66, την 66η επέτειο της απελευθέρωσης των κρατουμένων στο στρατόπεδο του Auschwitz. Σήμερα κλείνουν 66 χρόνια. Επίσης δημιουργήσαμε ένα φόρουμ που, όπου συμμετέχουν όλοι οι πρώην πρόεδροι του Ευρωκοινοβουλίου και έχουμε μέλη αυτού του φόρουμ εδώ, παρόντες στην αίθουσα, που δρούν εξ και για την πρωτοβουλία αγορά, που αποτελεί να παράγοντα, ένα φορέα σύνδεσης για όλες τις πρωτοβουλίες. Και γι' αυτό η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι τόσο σημαντική, διότι συμπεριλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες των πολιτών. Πριν από ένα χρόνο, μάλιστα, δημιουργήσαμε και ένα φόρουμ για την ελευθερία των Ευρωπαίων. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, ασχολούνται με την πρωτοβουλία αυτή. Και πάλι να ευχαριστήσω τους ε, αντιπροέδρους Ρούτσεκ και Ντουγάν και όλους όσους συνέβαλαν ώστε να είμαστε σήμερα όλοι συγκεντρωμένοι εδώ. Τέλος, μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. διανύουμε μια περίοδο κρίσης. Ο αριθμός των φτωχών ανθρώπων αυξάνεται σε περίοδους κρίσης. Περισσότερος κόσμος ε, φτωχός σημαίνει περισσότερα κοινωνικά προβλήματα και αυτό με τη σειρά του επιφέρει ε, περισσότερα προβλήματα ανάμεσα στα έθνη. θα πρέπει να θυμηθούμε μια άλλη κρίση την οποία διανύσαμε κατά την περίοδο του 1928 με 1931. Ε, τεράστια ανεργία και φτώχεια και ξέρουμε σε τι καταλήξαμε τότε. Θα πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν μας και να εξασφαλίσουμε ότι αυτή τη φορά θα ακολουθήσουμε διαφορετικό δρόμο. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει αυτή την πρωτοβουλία αγορά. Σας εύχομαι καρποφόρα συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την αρχική σας παρέμβαση και τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Λάσλο Άντορ, τον Επιτροπό Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Συμπερίληψης. Δηλαδή ασχολείται με τα ζητήματα της φτώχειας και της καταπολέμησής της. Να αναφέρω επίσης πως ο κύριος Επίτροπος θα πρέπει να φύγει μετά την ε, ομιλία του. να σημαίνει αυτό πως είναι αγενής. Όπως ξέρετε οι Επίτροποι έχουν πολλές υποχρεώσεις. Οπότε ζητά συγγνώμη των προτέρων και ε, ζητώ και εγώ συγγνώμη. Πρέπει να αποχωρήσει αμέσως μετά την ομιλία του. Κύριε Επίτροπε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μεγάλη ευχαρίστηση για εμένα να είμαι εδώ πέρα στην τρίτη αγορά πολιτών που οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Είναι ένα μεγάλο παράδειγμα συμμετοχικής δημοκρατίας και προσωπικά είναι τιμή μου να συμμετέχω. Όπως είπε και ο πρόεδρος Μπούζεκ, στην εισαγωγή του η σημερινή αγορά λαμβάνει χώρα μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και μας δίνει μια πραγματική ευκαιρία να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε μαζί και να ε, μπορέσουμε να βγούμε ένα δίκαιο και αηφόρο τρόπο από την κρίση. Υποστηρίζοντας την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των φτωχών, είναι βασικός ε, στόχος της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και θεωρώ πως το ευρωπαϊκό έτος, ε, το σχετικό το 2010 δηλαδή, επέτυχε ένα σημαντικό βήμα. Συναντήθηκαν αρκετοί διαφορετικοί φορείς, ε, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω η σημερινή εκδήλωση να αποτελέσει άλλη μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Κυρίε και κύριοι, ενώ ξεκινάμε, έχουμε τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης των οικονομιών μας από την ε, πάρα πολύ ισχυρή αυτή η οικονομική κρίση. Εξακολουθούν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι σε ολόκληρη την Ήπειρο να νιώθουν τον αντίκτυπό της. Ε, τα στατιστικά στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Υπάρχουν 5 εκατομμύρια περισσότεροι άνεργοι από την αρχή της κρίσης και πολλά περισσότερα νοικοκυριά έχουν δει το εισόδημά τους να πέφτει πάνω από ένα στους πέντε νέους Ευρωπαίους δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες μακροχρόνιου αποκλεισμού. Και πάνω από 80 εκατομμύρια ζουν υπό κίνδυνο φτώχειας. Βεβαίως πάρα πολλά. Το μεγάλο βάρος βέβαια το φέρνουν τα κράτη-μέλη, μιλάμε για τα στήματα κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης και στέγασης. Όμως ξέρουμε πως υπάρχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση Τρία τέταρτα των πολιτών μας, ακριβώς 74% στις δημοσκοπήσεις πιστεύουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει. Σύμφωνα με τα καετή στρατηγική μας για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο που λέγεται στρατηγική 2020, για πρώτη φορά η Κομισιόν πρότεινε συγκεκριμένο αριθμητικό στόχο για τη φτώχεια. Συμφώνησαν λοιπόν πως 20 ε, εκατομμύρια τουλάχιστον Ευρωπαίοι θα έχουν ξεφύγει από τη φτώχεια μέχρι το 2020. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο τα κράτη-μέλη πρέπει να θέσουν δικά τους φιλόδοξα εθνικά προγράμματα και στόχους θα αντικατοπτρίζουν την κατάσταση κάθε χώρας. Κυρίε και κύριοι, για να στηρίξουμε τις προσπάθειες ε, και την πρόοδο προς αυτό τον κύριο στόχο, πέρσι 16 Δεκεμβρίου η Κομισιόν υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Στόχο έχει να δημιουργήσει μια κοινή δέσμευση για δράση μεταξύ κρατών μελών, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και όλων των διαφερομένων και σκοπεύει να αυξήσει τον συντονισμό μεταξύ πολλών εταίρων στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και προωθεί ιδέες για καινοτομία και βελτιώσεις μπορούν να μας βοηθήσουν όλους πιο αποτελεσματικά με το να εστιάζουμε τους πόρους εκεί που έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, τι προτείνουμε. Πρώτα απ' όλα η πλατφόρμα προτείνει δράσεις σε ολόκληρο το φάσμα της πολιτικής πέρα από τις παραδοσιακές ε, πολιτικές. Συμπεριλαμβάνει παραδείγματος χάρη τον ενεργή ένταξη αυτών που δεν είναι στην ε, αγορά εργασία στην αντιμετώπιση τη παιδική φτώχεια το να γίνουν οι υπηρεσίε κοινωνικές πιο αποτελεσματικές ή να ανταποκρίνονται στις ε, νέες ανάγκες, συνένταξη μειονοτικών ομάδων όπως η να ανταποκρινονται στις νεες αναγκες ένταξη μειονοτικων ομαδων όπω η ρωμα και τέλο. Ε, ε, αντιμετώπιση του οικονομικού αποκλεισμού και τη ενεργειακή φτώχεια. Τέλο, προωθούμε την καινοτομία στην κοινωνική πολιτική για να μπορέσουμε να βρούμε φτηνές αποτελεσματικέ λύσεις για τον εξυγχρονισμό των κοινωνικών πολιτικών. Η Κομισιόν θέλει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν καινοτομία που θα βασίζεται σε στοιχεία για να αξιολογήσει τι νέε προτάσει. Τρίτον, η πλατφόρμα έχει προτάσει για το πώ θα αξιοποιηθούν καλύτερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια ω προ το αποτέλεσμα του. Παραδείγματο χάρη, το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 για να παίξει τον ρόλο του στη μείωση της φτώχειας. Και τέλος, η πλατφόρμα προβλέπει διευρυμένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και θα ενισχύσει επίσης το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας. Είμαι πεπισμένος πως η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της στόχες και του κοινωνικού αποκλεισμού θα μας βοηθήσει να βρούμε καινοτόμες ε, και διαρκείς ε, και οικονομικές λύσεις για τη φτώχεια στην Ευρώπη. Όπως σας είπα, οι Ρωμά επίσης αποτελούν αντικείμενο του ενδιαφέροντος μας. Επίσης, η πλατφόρμα αναφέρεται στους Ρώμα, που είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όμως είναι μια από τις ομάδες που είναι πιο κοινωνικά αποκλεισμένες. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι Ρωμά έχουν πάρα πολλά μεγάλα επίπεδα ηλικής στέρησης, ε, ανεργίας, μεγάλα και συχνά αυξανόμενα χάσματα στην εκπαίδευση, πάρα πολύ μεγάλες προκαταλήψεις και διακριτική μεταχείριση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολύπλοκα και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση που σημαίνει πως θα πρέπει να δούμε συνολικά το πού μεγαλώνει η Ρώμα μέχρι τη συμμετοχή του στην οικονομία και την κοινωνία. Το Σεπτέμβριο του 2010 η Κομισιόν δημιούργησε μια εσωτερική ομάδα δράσης για να αξιολογήσει πώς χρησιμοποιούν τα κονδύλια τα κράτη-μέλη και την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση στο Ρωμά. Τον Απρίλιο σκοπεύουμε να εξετάσουμε το έργο αυτής της ομάδας εργασίας ε, καθώς ε, και το τι είχε γίνει μέχρι το 2009 για να παρουσιάσουμε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Το πανευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο θα αξιολογήσει την χρήση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων και θα κάνει προτάσεις για πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την καταπολέμηση του αποκλεισμού των Ρωμά. Επιπλέον, το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα προσπαθήσει να διασφαλίσει καλύτερη επιτήρηση και στήριξη εθνικών και ευρωπαϊκών προσπαθειών προς αυτήν την κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, πραγματική πρόοδος για την καταπολέμηση της φτώχειας θα επιτευχθεί μόνο με την εμπλοκή όλων των διαφερομένων σε όλα τα επίπεδα. Εθνικό, τοπικό και ευρωπαϊκό η Κομισιόν θα συνεργαστεί με άλλα θεσμικά όργανα και φορείς για να μεταμορφωθεί αυτή η πλατφόρμα σε ένα ε, ευρύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο που θα λαμβάνει η χώρα τον ε, Οκτώβριο για να κάνουμε ένα απολογισμό της προόδου. Θα ε, βλέπουμε πώς έχουν εφαρμοστεί οι δραστηριότητές μας και βεβαίω να υποβάλουμε προτάσεις για τη μελλοντική δράση κατά πολέμηση της φτώχειας πρέπει να αποτελέσει μέρος της συνολικής στρατηγικής ανάκαμψης. Δεν είναι μόνο ηθικό καθήκον, αλλά και οικονομική αναγκαιότητα. Αναμένω λοιπόν τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους ενδιαφερομένους ΜΚΟ και τους ανθρώπους που ζουν στη φτώχεια για να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε σχέση με τους λόγους που εκφωνούν και θα ζητήσω παρακαλώ έλα παρακαλώ από το βήμα είχε δημιουργηθεί στην Γαλλία στη στην Γαλλία πριν από τέσσερα χρόνια και συναπατήστε από εθελοντές και άστεγους που έχουν συνενωθεί σε ένα κοινό εγχείρημα του να συμμεριστούν και να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα την περίοδο αυτή της έντονης κρίσης και της έκφρασης αλληλεγγύης. Σας ευχαριστούμε πολύ στα γαλλικά και στα αγγλικά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την χοροδία και το βράδυ μαζί μας στο δείπνο της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής και φυσικά και αύριο κατά τη διάρκεια της ορομέλειας της έναρξης της και επιτρέψτε μου να προαναγγείλω τον επόμενο αγόριτη, ο κύριος Πέτερ Γιώκες που είναι ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Η πρέσβης, θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος της, Ευρωπαϊκής, της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει την ανακυκλούμενη Προεδρία για έξι μήνες η Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι προεδρεύει σε αυτό το Συμβούλιο. Έχει τον λόγο κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, φυσικά μετά από αυτή την ε, εκτέλεση αυτών των τραγουδιών, αυτή την ερμηνεία δεν είναι εύκολο μετά από αυτά τα τραγούδια να επιστρέψει κανείς σε ένα καθαρά πολιτικό και θεσμικό επίπεδο στις διεργασίες και στην προσέγγιση την θεσμική. Πώς και πού μπορούμε να εντάξουμε και να επικεντρώσουμε τον αγώνα κατά της στόχια στις γενικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τις επιπτώσεις της τεράστιας αυτής κρίσης. Όμως ωστόσο θεωρώ ότι Υπάρχει κάποιος αξιόλογος, ε, κάποιος τόπος που, στον οποίο ένα κέντρο στο οποίο μπορούμε να επικεντρωθούμε για να διεξαγάγουμε αυτόν τον αγώνα με θετικό τρόπο. Και μια και αυτό είναι ο κινητήριος, ε, η κινητήρια δύναμη όσον αφορά κατά την ίδια τη διάρκεια της ε, Προεδρίας της Ουγγαρίας στο Συμβούλιο και ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι χρήσιμο ιδιαίτερα για εκείνους που θα συμμετάσχουν σε αυτό τον ενεργό διάλογο με τα θεσμικά όργανα και την κοινωνία των πολιτών με αυτόν τον τρόπο να επικεντρωθούν ώστε αυτός ο αγώνας να είναι αποτελεσματικός ε, για την επίτευξη της στρατηγικής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρώπη του 2020. Να σας διασφαλίσω επίσης ότι η Ουγγρική Προεδρία έχει πολύ ανοιχτό πνεύμα σε αυτό το πεδίο για ένα διάλογο μαζί σας. Η αφετηρία είναι ότι θα εναρμονίσουμε και θα συντονίσουμε τις προσεγγίσεις μας. Πώς αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική θα διαμορφωθεί, πώς πρέπει να διαμορφωθεί. Υποθέτω ότι το σημείο κίνησης είναι το εξής. Η Ευρώπη που χρειάζεται χρόνο για να αφομοιώσει και να χωνέψει ότι βρισκόμαστε μέσα στο επίκεντρο, στη μέση μιας τεράστιας ε, πελώριας κρίσης που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμιά άλλη κρίση με τις κρίσεις που είχαμε στο παρελθόν. Και κάτι δεύτερο ακόμα, ότι για να διεξέλθουμε, να διαφύγουμε από αυτή την κρίση χρειαζόμαστε ε, νέα μέσα και εργαλεία. Αυτή είναι ουσιαστικά η ανάλυση και οι συνιστώσεις της. Ε και για την ε, εκπόνηση μια ε, προσέγγιση ενό οράματο πώς από πλευρά Ευρώπη πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον μα, Δηλαδή, αυτή είναι ακριβώ η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Και αυτή η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, σε αυτήν η καταπολέμηση τη φτώχεια διαδραματίζει ένα θεμελιώδη ρόλο. Γιατί είναι φυσικά μία, ένας από τους κύριους άξονες, ε, ένας στόχος που πρέπει να πετύχουμε μέχρι το 2020, να μπορέσουμε να αυξήσουμε ε, κατά 30% τον αριθμό εκείνων των πολιτών ε, που θα πρέπει να διαφύγουν από το κατόφλι της στόχιας και να μπορέσουν να ζήσουν σε ευημερία. Το θέμα είναι ότι δεν είναι δύσκολο να εκπονήσει κανεί κάποια τέτοια οράματα και προσεγγίσεις. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να πετύχει να προσεγγίσει τέτοιου είδου στόχου. Και κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, εφέτο, θα πρέπει να καταρτιστεί αυτή η πορεία και όλα τα μέσα και εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ε, βρίσκονται για παράδειγμα όπως η ε, τροποποίηση της συνθήκης ε, η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσης για την σταθεροποίηση της οικονομίας με, την ευρωορολογία κάνοντας λόγο για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Μα περί τίνος πρόκειται εδώ ουσιαστικά. Είναι η δημιουργία μιας νομικής βάσης ουσιαστικά για να δημιουργηθούν τα αναγκαία πλαίσια ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον η Ευρώπη να εμπλακεί σε μια τέτοια κρίση. Από την άλλη όμως πλευρά μην ξεχνάμε σίγουρα ότι αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και εξυγίανση δεν επαρκεί για να καταπολεμηθούν όλα τα αρνητικά φαινόμενα στις κοινωνίες μας. Και γι' αυτό πρέπει να αντιληφθούμε και κάτι άλλο, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η κρίση δημιούργησε, προκάλεσε κάποιες επιπτώσεις που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ότι δεν μπορούμε μόνο να επικεντρωνόμαστε σε προκλήσεις ή προβλήματα τα οποία είχαμε ήδη στο παρελθόν, για παράδειγμα στο τομέα, στο πεδίο της φτώχειας. Αυτή η κρίση δημιούργησε απόλυτα νέα φαινόμενα, νέες μορφές φτώχειας. Τούτων λεχθέντων λοιπόν ποια πρέπει να είναι η προσέγγιση, οι διεργασίες, ποιες πρέπει να είναι αυτές. Τώρα λοιπόν, μετά από τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης, μετά από τη δημιουργία όλων των πολιτικών και νομικών μέσων και εργαλείων, πρέπει να ειναι η προσεγγιση οι διεργασιες ποιε πρεπει να ειναι αυτες τωρα λοιπον μετα απο τη σταθεροποιηση της ευρωζωνης μετα απο τη δημιουργια ολων των πολιτικων και νομικων μεσων και εργαλειων πρεπει να επικεντρωθουμε στην αηφόρο ανάπτυξη στην ανάπτυξη που θα είναι φιλική για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και επίσης εκείνα τα μέρη, τα τμήματα της κοινωνίας μας που δεν μπορούσαν μόνα τους να ε, διαφύγουν από τη φτώχεια και από τις, ε, την πιεστική αυτή κατάσταση που δημιούργησε η κρίση να βοηθηθούν και να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, ένα δομημένο, διαρθρωμένο διάλογο σε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να δράσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγρική Προεδρία στοχεύει να έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για αυτά τα θέματα με το, ε, ήδη τον Μάρτιο. Αυτό είναι η μία πτυχή. Μα, ε, δεύτερη πτυχή, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική ώστε να στεφτεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα της Ευρώπης του 2020. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η δράση θα βαίνει εκ παραλίλου και θα εξελίσσεται σε δύο επίπεδα. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο αφενός και στο εθνικό επίπεδο αφετέρου. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν θα υιοθετήσουμε με το Συμβούλιο του Μαρτίου τις αντίστοιχες κατευθυντήρες γραμμές ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ω σύνολο να μπορέσει να κινητοποιηθεί προ μια ενιαία κατεύθυνση. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να γνωρίζει κανεί ότι με αυτή τη βάση τον Απρίλιο τα 27 κράτη-μέλη θα κάνουν το εξή. Θα πρέπει να υποβάλουν τα εθνικά προγράμματα αναθεώρηση και μεταρρύθμιση και μέσα σε αυτά τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν συγκεκριμένες δεσμευτικές ενδείξεις και να αναλάβουν συγκεκριμένη πορεία που θα δείχνουν πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί από τους κυριότερους στόχους. Και ένας από τους πέντε κυριότερους στόχους είναι ακριβώς η καταπολέμηση της φτώχειας. Και εδώ ακριβώ πρέπει να δεσμευτούμε με ιδιαίτερα στεναρό και αποτελεσματικό τρόπο και να σχεδιαστούν τα εθνικά μέτρα πολιτική ώστε να επιτευχθεί αυτό ο στόχο, να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί τελικά. Επιτρέψτε μου στη συνέχεια να επανέλθω, να έρθω τώρα σε ένα άλλο στοιχείο, το οποίο θα διαδραματίσει, ήδη διαδραματίζει σε έναν ουσιώδη ρόλο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και του προγράμματός μας ε, ως Ουγγρικής Προεδρίας. Αυτό είναι η στρατηγική για τους Ρωμά, για τους Τσιγκάνους. Όχι μόνο οι Τσιγκάνοι υφίστανται τα δεινά και τις επιπτώσεις της φτώχειας, αλλά ίσως και αυτό είναι, είναι η πιο ευάλωτη όλου, από όλο τον πληθυσμό μας η Τσιγκάνη, η πιο ευάλωτη ομάδα. Και είναι στεναρός μας, στεναρή μας πρόθεση με κάθε αποφασιστικότητα να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις στρατηγικές για τους τσιγκάνους ε, κατά τα τέλη της Ουγγρικής μας Προεδρίας. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένουμε να δημοσιοποιηθεί στις αρχές Απριλίου σε αυτό το συγκεκριμένο πεδίο θα έχουμε ένα διαρθρωμένο, δομημένο διάλογο και πολιτική που θα ακολουθηθεί στις διαφορετικές, στα διαφορετικά επίπεδα από πλευρά του Συμβουλίου. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα για τους τσιγκάν, των τσιγκάνων με την φτώχεια, την ε, ε, έλλειψη παιδείας και εκπαίδευσης της ανεργίας θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Βλέπετε υψηλό βαθμό συνέργειας σε σχέση με αυτές τις δράσεις για, τη, για τους στόχους της Ευρώπης 2020. Και στη συνέχεια είναι στεναρή μας ε, αμετακίνητη πολιτική μας απόφαση ως στόχος να ξεκινήσουμε και να έχουμε αυτή τη στρατηγική που θα εγκριθεί τον Ιούνιο από πλευρά τη Συνόδου Κορυφή του Συμβουλίου για την πολιτική για του Τσιγκάνου. Βλέπετε λοιπόν, εδώ υπάρχει μια δέσμη πολιτικών μέτρων και εργαλείων με υψηλέ φιλοδοξίε. Η Ουγγρική Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σα προσκαλεί να ξεκινήσει αυτό ο διάλογο και να εμπλακείτε σε αυτόν ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό ο στόχο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη και θα ελπίζουμε και θα ευχόμαστε κάθε επιτυχία ευχόμαστε στην Ουγγρική Προεδρία για αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Our next speaker is Mr. Ο επόμενος αγορητής Στέφαν Νίλσεν, πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με άλλα λόγια εκπρόσωπος της ε, διαφρομένης οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό στο μέλλον. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά και θα συνεργαζόμαστε και στο μέλλον με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή. Στο Ευρωκοινοβούλιο είμαστε οι αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών από 27 κράτη-μέλη εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια πολίτες. Αν θέλουμε όμως να στεφτούν με επιτυχία τα εγχειρήματά μας, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, επίσης και στον στόχο της καταπολέμησης της φτώχειας και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, πρέπει και θέλουμε να συνεργαστούμε και με άλλα θεσμικά όργανα και φυσικά η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι ένα από τα πιο σημαντικά από αυτά τα θεσμικά όργανα. Λοιπόν, τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Νίλσον, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να πω στη δική μου γλώσσα στα ειδικά κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό σε σχέση με την παρέμβαση του Πρόεδρου που έγινε στα αγγλικά. Μετά θα συνεχίσω στα αγγλικά και εγώ, διότι θα ήθελα φυσικά να διασφαλίσω ότι άμεσα θα μπορώ να στραφώ σε εσάς και να με κατανοήσετε από πρώτο χέρι. Λοιπόν, συμφωνώ. Ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτή η χοροδία. Είναι ένα καλό παράδειγμα ότι η μουσική διασυνοριακά γίνεται κατανοητή από όλους τους ανθρώπους. Πέρα από γλωσσικούς φραγμούς η μουσική, η μελωδία είναι μια διεθνής γλώσσα. Ευχαριστώ θερμά για αυτό που ήταν πολύ θετικό λοιπόν και μα συγκίνησε. Δεύτερον, θα ήθελα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πω ότι Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τις ε, πρωτοβουλίες ε, σεβόμαστε το Ευρωκοινοβούλιο και θεωρούμε ότι είναι ένα όργανο που λαμβάνει αποφάσεις ε, μεγάλης εμβέλειας μεγάλης εμβέλειας αποφάσεις και φυσικά νομοθετεί, συνομοθετεί ως συνομοθέτης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή λοιπόν έχει 374 μέλη και έχουμε και μέλη που εκπροσωπούν όλους τους τομείς ε, και από όλες τις χώρες ε, και εκπροσωπούν έτσι οι πολίτες και ελπίζουμε ότι μπορεί με αυτή την απήχηση να καλύπτονται οι ανάγκες των πολιτών και ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω να πω ότι έχουμε ένα κοινό στόχο ενώπιόν μας σε αυτή μας την κοινή συνεδρίαση. Δεν είμαστε ο ένας κάτω από τον άλλο, υφιστάμενος ο ένας του άλλου. Αντίθετα είμαστε ισότιμοι και εργαζόμαστε δίπλα-δίπλα ο ένας, δίπλα στον άλλο σε, ένα κοινό, σε μια κοινή προσπάθεια που προσπαθούμε να εκδοκιμήσει. Χαίρομαι που μπορώ εδώ σε σχέση με την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή να παρέμβω. Είμαστε ένα όργανο το οποίο βρίσκεται διαρκώς σε διαβουλεύσεις και συζητήσεις όπως και στην αγορά των πολιτών. Συζητούμε με τους εκπροσώπους των πολιτών, καταναλωτές, εκπροσώπους οργανώσεων για τα δικαιώματα των πολιτών, ε, υπέρμαχους των δικαιωμάτων αυτών και συνεργαζόμαστε με δραστήριο τρόπο να μπορέσουν να, πετύχουν, να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Χαίρομαι για το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ συνενωμένοι και ότι έχουμε και τις ομάδες που εκπροσωπούνται σε εμάς οι τρεις ομάδες που διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα ήθελα τούτων λεχθέντων Ιζαμπέρ να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία Όλοι είμαστε πεισμένοι ακράδαντα για το γεγονός ότι αυτή η σύγκληση της αγοράς αυτής είναι μία ακόμα απόδειξη, χειροπιαστή απόδειξη για την καλή συνεργασία που έχουμε. Το μήνυμα που κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, κατά τη διάρκεια 4,5 ετών της Προεδρίας δηλαδή στην κοινωνική και κοινωνική, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή το μήνυμα είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη της αηφορίας, της ανάπτυξης και της ευημερία. Νομίζω ότι αν, τα, αν καταβάλουμε προσπάθειες από κοινού θα τα καταφέρουμε η ε, σύνοδος αυτή της αγοράς σε εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά με ένα σωστό τρόπο και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που προσφέρονται. Έχει δικαίωμα κάθε ένας από εμά να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε και με βάση τη νέα συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας, είναι ακόμα πιο σημαντικό Όλοι οι πολίτες θα μπορούν έτσι με αυτόν τον τρόπο να συμμετέχουν στις ε, διαδικασίες της ε, ε, που βρίσκονται υπό εξέλιξη και να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τις διάφορες μορφές της φτώχειας που είναι ένας, ένα περίπλοκο εγχείρημα ιδιαίτερα τώρα όταν η μέγιστη μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται ακριβώς προς τα ευρωπαϊκά οικονομικά ζητήματα προς την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι κοινωνικές προκλήσεις ε, που ε, υποδαβλίστηκαν και ε, δημιουργήθηκαν από αυτή την κρίση πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο ότι θα εγγραφούν σε υψηλό επίπεδο προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη όπως το κάνουμε εμείς εξάλλου εδώ σε αυτή την αγορά. Αυτό το φόρουμ λοιπόν έχει στόχο να ισορροπήσει, να εξισορροπήσει τα θέματα στην πολιτική συζήτηση και προσέγγιση. Τρίτον, επειδή είδα ακριβώς το ενδιαφέρον που έχετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξει μια ευρύτερη δυνατόν εκπροσώπηση και συμμετοχή στις συζητήσεις της αγοράς της κοινωνίας των πολιτών και ε, συνεργαστήκαμε πολύ στενά για να προετοιμαστεί αυτή η προσέγγιση και εμείς από πλευράς μας θέλουμε να διασφαλιστεί ότι η κοινωνία των πολιτών όσο το δυνατόν σε ευρύτερο μεγαλύτερο βαθμό θα εκπροσωπηθεί ρόλος είναι να υποστηριχθεί ακριβώς ο διάλογος με τις οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε ότι θετικά θα εκπροσωπούνται όπως ε, συνάδει με αυτές και ότι θα συνεισφέρουν έτσι με αυτόν τον τρόπο στις εργασίες αυτού του φόρουμ. Έτσι λοιπόν σας ευχαριστούμε πολύ για το γεγονός ε, ότι είσαστε εδώ και βρισκόμαστε όλοι εδώ. Πρέπει να βρούμε πιστεύω ποιες λύσεις συνεισφέρουν στην αηφορία ώστε να διασφαλιστεί μια σωστή ένταξη και υποστήριξη ε, με ολοκληρωμένο τρόπο των ομάδων που αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα στην ε, κοινωνία μας. Αν τα καταφέρουμε και εδώ θα θέλουμε, να πούμε ότι πραγματικά αν καταβάλουμε τις προσπάθειες που πρέπει μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τότε οι φτωχοί άνθρωποι, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι και που αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους υπερήλικες, άτομα με μειονεξίες, ειδικέ ανάγκες, μετανάστες, Ρωμά Τσιγκάνοι και άλλες μειονότητες, ευάλωτες ομάδες. Θα είναι σε θέση να δουν ότι οι συνθήκες διαβίωσης τους μπορούν να βελτιωθούν. Η φιλοδοξία λοιπόν της, ευρωπαϊκής, της πολιτικής ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειωθεί ε, το εύρος της φτώχειας και να μειωθεί ο αριθμός κατά 20 εκατομμύρια πολίτες, των φτωχών πολιτών δηλαδή, να μειωθεί ο αριθμός κατά 20 εκατομμύρια μέχρι το 2020, αν είμαστε πραγματικά φιλόδοξοι και καταβάλουμε προσπάθειες, δεν είναι κάτι το ανέφικτο αυτό. Θεωρούμε όμως από την άλλη πλευρά ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις και με πλήρη υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και πλήρη εμπλοκή όλων μας ε, θα πρέπει να οδηγήσουν σε αυτές τις, ε, στην ανάπτυξη των προσπαθειών. Επίσης, ε, σε σχέση με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είμαι βέβαιος ότι όσοι είναι παρόντες και παρούσες σε αυτή την ε, σύγκληση, σε αυτή την ε, σύνοδο αγοράς, θα συνεισφέρουν και θα δώσουν τις συμβουλές τους και τις γνώμες τους γνωμοδοτώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να γίνει. Μία από τις σημαντικές συστάσεις μας είναι ότι οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ολοκλήρωσης πρέπει να είναι στενά συνδυασμένες με τις ε, πολιτικές που θα ακολουθηθούν για την ε, ανάπτυξη της οικονομίας μας ε, και να μπορέσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να ενταχθούν ενεργά οι γνώμες μας και να δούμε πώς μπορεί η Ευρώπη να ξεφύγει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το 2011 θα συνεργαστούμε για την ένταξη, την κοινωνική ένταξη των τσιγκάνων, των μεταναστών και θα αντιμετωπίσουμε το θέμα, το πρόβλημα των αστέγων και του κοινωνικού αποκλεισμού θα επικεντρώσουμε τη δουλειά μας σε τρία οριζόντια εγκάρσια θέματα ως προτεραιότητες. Διάλογο και συμμετοχή, αηφορία και ανάπτυξη, αλληλεγγύη και ανάπτυξη. Και μέσα σε αυτό το συνολικό πλαίσιο κοινών ευθυνών και κοινή ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας για την αντιμετώπιση, την μείωση του αριθμού των φτωχών μέχρι το 2015. Θα έχουμε και την διάσκεψη για την ασφάλεια ε, των τροφίμων. Αποκινούμε τον ε, ΦΑΟ, ε, τον Οργανισμό Τροφίμων και επισητισμού των Ηνωμένων Εθνών καθώς επίσης και υπό την σύνοδο της G20 διότι έχει εγγραφεί το θέμα αυτό για τον Ιούνιο στην ημερήσια διάταξη της συνόδου αυτής. Πρέπει να πω ότι προσβλέπω ιδιαίτερα να ακούσω και τις απόψεις σας και να μάθω από τις απόψεις σας και ελπίζω ότι θα έχουμε μια ζωντανή συζήτηση που θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε αυτά τα workshops, σε αυτά τα σεμινάρια. Η δική σας πείρα και και η γνώση σας ε, από κοινού ε, με την ε, στεναρή δέσμευση και τις προσπάθειες που ε, καταβάλλονται ελπίζω ότι θα δώσουν δυνατότητες να υπάρξουν λύσεις με, αηφόρο, με αηφορία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δράτω με ήδη τώρα της ευκαιρίας να σας προσκαλέσω στην συνάντηση που θα έχουμε στο κτίριο αυτό για ένα ποτό και Ελπίζω ότι θα έχουμε με αυτόν τον τρόπο ένα θετικό πλαίσιο συνεργασίας. Καμιά φορά συναντά κάποιους, κα, κανείς που δεν τους γνωρίζει και μπορεί να είναι ένα, μια θετική έκβαση κάτι τέτοιο, μια τέτοια επαφή που δίνει την δυνατότητα να γνωρίσει ο ένας τον άλλο καλύτερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν καλά, πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να προσφωνήσω το φόρουμ την αγορά. Θα συμμετάσχουμε όπως συμμετέχουμε και ελπίζω ότι η έκβαση θα είναι για όλους θετική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε Στέφαν, ευχαριστούμε κύριε Νίλσεν και για να στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα πρέπει να αναπτύξουμε στρατηγικέ συνέργειες σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και στο επίπεδο των κρατών μελών και στο επίπεδο των περιφερειών. Και γι' αυτό τον λόγο προσκαλέσαμε ακριβώς και την κυρία Μπρεσό, πρόεδρο της Επιτροπής ε, των περιφερειών για να μας διαφωτίσει τι μπορεί να γίνει και στο επίπεδο της Επιτροπής των Περιφερειών. Δυστυχώς άκουσα ότι υπήρχαν πρόβλημα μεταφοράς και έτσι δεν μπόρεσε έγκαιρα να είναι παρούσα εδώ. Και έτσι θα δώσουμε 10 λεπτά ή ένα τέταρτο ακόμα μέχρι να προσέθει. Εν τω μεταξύ θα γίνουν κάποιες ε, τεχνικές, ε, τεχνικής μορφής και θα δούμε αν εν τω μεταξύ θα καταφέρει να φτάσει εδώ πριν από το γεύμα. Λοιπόν, μετά από αυτή τη σημερινή συνεδρίαση αυτού του πρωινού θα έχουμε γεύμα στο χώρο Γεχούντι Μενουχίν που βρίσκεται στον πρώτο όροφο εδώ αυτού του κτηρίου. Απλά θα πρέπει να κατέβετε από τα, από τα σκαλιά ή να πάρετε τον ανελκυστήρα και να πάτε στο πρώτο όροφο. Στις 2.30 θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας σε ομάδες εργασίας, workshops, στο κτίριο Αλτιέρο Σπινέλη. Είναι το κτίριο στο οποίο φτάνετε όταν περάσετε αυτή τη γέφυρα ε, ε, το πρώτο workshop για τις νέες μορφές φτώχεια στην αίθουσα 3G3 πάλι στον τρίτο όροφο του ορόφου Αλτιέρο ε, Σπινέλη. Δεν θα πρέπει ούτε να ανέβετε ούτε να κατέβετε. Είναι στον τρίτο όροφο απέναντι. Μετά όσον αφορά τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη στο 3G2 ως αίθουσα κοντινή αίθουσα και το τρίτο σεμινάριο για το, τη μορφή της κοινωνίας που θέλουμε να ε, δημιουργηθεί θα είναι στο 1G3, στο πρώτο όροφο το G3 και για την συμμετοχή στην συνενετική διάσκεψη στο 5G3, δηλαδή στο πέμπτο όροφο στο G3 στον χώρο που ήδη υπήρξε συνάντηση εχθές. Θα εργαστείτε υπό την πρωτοκαθεδρία των αντίστοιχων συντονιστών που θα αναλάβουν την Προεδρία και ελπίζουμε ότι τα συμπεράσματα των, διαφορετικών, των διαφόρων εισηγητών των ομάδων εργασίας και σεμιναρίων θα τα ακούσουμε αύριο το πρωί σε αυτή την αίθουσα 9 η ώρα το πρωί. Θα ακολουθηθεί ε, από μια συζήτηση στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι συμμετέχουν και ελπίζω ότι αθρώα θα είναι η συμμετοχή σας στη συμμετοχή σε, σε αυτή τη συζήτηση ακριβώς διότι στόχος δεν είναι μόνο να ακούσουμε σήμερα και αύριο τους λόγους που θα εκφωνήσουν οι διάφοροι αρμόδιοι, αλλά να εκφράσετε εσείς οι ίδιοι προσωπικά τις απόψεις σας ε, και τα ε, αισθήματά, το τι αισθάνεστε. Και για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση θα ζητηθεί να καταχωρήσετε τα ονόματά σας σε ένα δελτίο που θα βρείτε εκεί στα τραπέζια δελτία συμμετοχής με τα στοιχεία, το όνομά σας και τα στοιχεία σας. Μπορείτε να τα, δείτε, να τα δώσετε ή στη γραμματεία της αγοράς ή στους κλητήρες ώστε να μπορέσουν να διαβιβαστούν στους αρμόδιους. Έτσι θα γνωρίζει και ο πρόεδρος και το όνομά σας και το ποιοι είσαστε και θα γνωρίζουν έτσι και οι συνάδελφοι ε, τα σχετικά με εσάς. Μια άλλη ανακοίνωση που αφορά το αποψινό δείπνο για τους ε, καταχωρημένους ε, συμμετέχοντες. Πρόσκληση στις 18 ε, και 45 στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής στην Οδό Μπελιάρ, στο επόμενο πιο κοντινό κτίριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να φτάσετε σε αυτό το κτίριο θα ζητούσα να κρατήσετε το badge που έχετε, την ταυτότητά σας, ώστε να μπορείτε να εισέλθετε εκεί. Διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα ασφάλειας και μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες για να γίνετε δεκτοί εκεί και να περάσετε στο κτίριο. Θα φύγουμε από εκεί από το κτίριο ε, του Κοινοβουλίου στις 6.30 και έτσι θα μπορέσετε όλοι από κοινού να πάτε με τη συνοδεία μας στο άλλο κτίριο και να είναι η μετάβασή σας πιο εύκολη. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, κάποια σχόλια, κάποιες απορίες που θα θέλατε να διατυπώσετε. Εσείς παρακαλώ, η κυρία στην τέταρτη σειρά. Θέλετε να πατήσετε το κουμπί του μικροφόνου εσείς στην τέταρτη σειρά, κυρία. Sorry. Με συγχωρείτε. Ναι, ανησύχησα που αναφερθήκατε στο πρόβλημα των Ρωμά. Δεν είναι πρόβλημα των Ρωμά. Οι άνθρωποι έχουν το πρόβλημα, όχι οι Ρωμά. Δεν θα λέγατε το εβραϊκό πρόβλημα, γιατί ξέρουμε που οδήγησε αυτό. Και πρέπει να ξανασκεφτείτε λίγο τη φρασιολογία σας. Thank you. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο αυτό. Κάποιος άλλος. Ο κύριος στην τέταρτη σειρά. Γεια σας, ε, Φιλίπ Προαγέ, Πρόεδρος της ε, Ευρώπης ε, των Φοιτητών. Σας ευχαριστώ για την διεξαγωγή αυτής της συνεδρίασης για τόσο λεπτό θέμα της φτώχειας, αν και λυπάμαι για τη φτώχεια της διάδοσης της εκδήλωσης αυτής πριν από λίγο ο πρόεδρος Μπούζικ είπε ότι η αγορά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ε, της ε, συμμετοχικής δημοκρατίας, όμως η φτώχεια είναι το ακριβώς αντίθετο, η ακριβώς αντίθετη απόδειξη της, ε, της συμμετοχικής δημοκρατίας. Πιστεύω ότι ναι, ο κοινωνικός τομέας δεν είναι αρμοδιότητα του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά περισσότερο αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί πραγματικά να πιστεύει ότι θα αντιδράσει με συγκεκριμένο και αποτελεσματικό τρόπο για να καταπολεμήσει τη φτώχεια ή θα μείνει απλά ένας ε, παρατηρητής της φτώχειας με μια προσέγγιση ε, οικονομική και όχι ε, λειτουργική και ανθρώπινη. Ευχαριστώ. Μάλκομ Ντάουρ λέγομαι και εκπροσωπώ την ΑΡΚΑ την Ευρωπαϊκή Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση, μια ένωση μη κυβερνητικών οργανώσεων από πολλούς τομείς, ε, μεταξύ των οποίων και ε, οργανώσεων που καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό στις περιοχές υπαίθρου. Σωστά καλέσατε τον Επίτροπο τον κύριο Έντορ, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα μέρη και τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των θεσμικών οργάνων που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη μοίρα των φτωχών και ευάλωτων. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι ο Επίτροπος ο κύριος Έντορ μαζί με τον κύριο Τσόλος και τον κύριο Χάν της ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Επίτροπο Αλίας ε, και ζήτησαν ε, η επόμενη προγραμματική περίοδος να έχει μια κοινή στρατηγική μεταξύ των πέντε κοινωνικών ταμείων, δηλαδή περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, ε, αλίας, για να δούμε το ζήτημα της πραγματικής ανάπτυξης όπως χρησιμοποιείται και στον τρίτο κόσμο κάτι το οποίο θα βοηθήσει μεταξύ άλλων τους φτωχού και τους ευάλωτους και εμείς στην ανακοίνωσή μας για την συζήτηση για την μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική. Έχουμε ευστήσει την προσοχή στις ανάγκες των φτωχών και ευαλώτων και το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν στα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης. Αποκινούμε τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και τα κοινωνικά και τα ζητήματα αλίας. Οπότε θα σας παρακαλούσα να διευρύνετε την συζήτησή σας από την αφετηρία που είναι βεβαίως ε, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων και να αναγνωρίσετε πως ε, πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές ε, επηρεάζουν τους φτωχούς και τους αποκλεισμένους. Ευχαριστώ. Πριν απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις θα δώσω και σε άλλους τον λόγο. Η κυρία στο 241. Μικαϊονίδου λέγομαι από την Ελλάδα Προέρχομαι από την ε, ελληνική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, που είναι η μεγαλύτερη γυναικεία οργάνωση της Ευρώπης. Είναι μια ε, ε, ομπρέλα οργανώσεων από όλα τα κράτη-μέλη και έχουν αντιπροσωπείες σε όλες τις χώρες. Ε, χαίρομαι που σήμερα ξαναβρίσκομαι εδώ γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτός ο θεσμός που άρχισε πριν από δύο χρόνια θα πρέπει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να ενδυναμωθεί. Θεωρώ ότι και η σημερινή συνάντηση όπως και οι προηγούμενες δύο είχαν αποτελέσματα. Απλώς πιστεύω ότι αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να επικεντρωθούν σε συμπεράσματα και σε κάποια πρακτικά μέτρα ώστε να μπορέσουν να περάσουν και στις χώρες. Η κοινωνία των πολιτών, στη χώρα μου για παράδειγμα, δεν έχει ακόμη ευαισθητοποιηθεί βάσει των συμπερασμάτων που έγιναν τις περασμένες χρονιές. Άρα θα έλεγα ότι χρειάζεται μια πιο, ε, σημαντική πολιτική ε, επικεντρωμένη στη διάδοση αυτού που γίνεται σήμερα εδώ. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό που ελέγχθη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δύναμη και αρμοδιότητες αλίμονο η φωνή των λαών να μην ακούγεται μέσα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι εκείνο που θα πρέπει να πιέσει να δώσει τη σημαντική όθηση στα θέματα τα κοινωνικά γιατί σήμερα στην ευρώπη που ζούμε στην ευρώπη της κρίσης η χώρα μου για παράδειγμα περνάει μια ανεπανάληπτη κρίση. δεν υπάρχει κανένα σημείο προς το παρόν το οποίο να δίνει ελπίδα στους φτωχότερους πολίτες. η δημοσιονομική προσαρμογή η οποία βεβαίως είναι αποτέλεσμα συμφωνίας αλλά μια συμφωνίας πάρα πολύ δύσκολης για το λαό πλήττει τους λιγότερο ευνοημένους. και πάνω απ' όλα θέλω να επικεντρώσω και το θέμα στις ε, γυναίκες που σήμερα στην Ελλάδα είναι εκείνες που πλήττονται έτσι και αλλιώς σε όλη την Ευρώπη, πλήττονται περισσότερο και κατά διπλάσιο τρόπο από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ενώ γυναίκες μεταξύ ανδρών δύο φορές παραπάνω είναι οι άνεργες γυναίκες και σήμερα στη χώρα και σε ολόκληρη την Ευρώπη οδηγούνται με έναν τρόπο ασφαλή στην ανεργία. Οι γυναίκες σήμερα δεν είναι μια ειδική κατηγορία. Είναι το μισό και παραπάνω του πληθυσμού αυτής της ενωμένης ευρώπης της ευρώπης αυτής που μας έδωσε οράματα και αυτής που πρέπει γρήγορα και υπάρχουν πολιτικές οι οποίες όμως ακόμη είναι στα επίπεδα πιστεύω του σχεδιασμού. απόδειξη επαναλαμβάνω μια χώρα που διέρχεται κρίση όπου σήμερα δημιουργούνται νέοι πολίτες που είναι πλέον μπαίνουν με ασφαλώς τη φτώχεια και πρώτα απ' όλα είναι οι νέοι και οι γυναίκες. Έχουμε διπλάσιους και τριπλάσιους αριθμούς και μακάρι αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας να είχε τα αποτελέσματα. Φοβάμαι ότι κάτω από αυτή την κρίση και αν δεν επικεντρωθούν οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως στο δημοσιονομικό όχι μόνο στο δημοσιονομικό αλλά στο κοινωνικό ζήτημα δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτή η κρίση και δεν είναι μόνο δημοσιονομική. Είναι κυρίως κοινωνική και είναι κρίμα η Ευρώπη στην οποία οικοδομήσαμε μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών να κινδυνεύσει για λόγους οι οποίοι οφείλονται σε καθαρά οικονομικούς, ε, ε, οικονομική αντιμετώπιση. Η παγκόσμια κοινότητα νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει σημασία πλέον στο ότι η ευρώπη είναι μια ανερχόμενη δύναμη η οποία δεν έχει μόνο οικονομικούς στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you. The gentleman 121. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εδώ και 25 χρόνια παρακολουθώ τους άστεγους στον ε, κεντρικό σταθμό. Ε, τις ομιλίες σας τις άκουσα, μιλήσατε για τους Ρωμά ή δεν ξέρω ποιους που έχουν ε, αυτοκίνητα και σπίτια, αλλά δεν μιλάτε για τους άστεγους. Και να σας πω ότι οι άστεγοι εξεκολουθούν να είναι στο δρόμο. Και να σας πω κάτι. Πάντοτε υπάρχει μια αρνητική εικόνα για τους αστέγους, αλλά οι πλούσιοι οι πλούσιοι δεν έχουν παρά μόνο μία σκέψη, την τσέπη του. Οι άστεγοι δεν έχουν παρά μόνο μία σκέψη, είναι η αγάπη των άλλων προς αυτούς. Ο κύριος το 235. Παγκύπρια οργάνωση μεγάλων οικογενειών ε, κάτω από την ομπρέλα της ΚΟΦΑΣΕ. Ε, δεν ακούμε να αναφέρεται καθόλου στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων οι πολυμελείς οικογένειες. Δεν αναφέρονται καθόλου. Ε, από την κρίση, με την κοινή λογική τουλάχιστον, μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε ότι πλήττονται κατά μαθηματική πρόοδο. Ε, γιατί το κατακεφαλήν εισόδημα της οικογένειας, μιας πολυμελούς οικογένειας, είναι πολύ πλέον χαμηλότερο από μια άλλη οικογένεια με ένα ή δύο παιδιά αυτές οι οικογένειες από την κρίση πλήττονται πολύ περισσότερο από όλες. Και αντίθετα, ε, σε βάθος χρόνου προσφέρουν πολύ περισσότερο από όλες τις άλλες οικογένειες, ε, όπως η δημογραφική ανέλυξη, το ακαθάριστο εισόδημα της χώρας και συνεπώς και η ευημερία της χώρας. Και μου φαίνεται ότι είναι άδικο να μην γίνεται μια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση και να μην αναφέρονται οι πολυμελείς οικογένειες μέσα στις ευάλωτες ομάδες. Ευχαριστώ. Thank you, gentlemen. Ευχαριστώ κύριο στο 202. Ε, <coughs> ε, ε. Ευχαριστώ, Μισελ Ρεκιέ. Δεν άκουσα να αναφέρεται σήμερα το πρωί η υπόθεση των ηλικιωμένων ανθρώπων που είναι εκατομμύρια στην Ευρώπη, πολλοί εξ αυτών βρίσκονται σε κατάσταση, κινδυνεύουν μάλλον από τη φτώχεια και άλλοι ε, μάλλον θα μπουν σε σειρέ των φτωχών λόγω των μηχανισμών μεταρρύθμισης των συντάξεων. Αν στις κατηγορίες που αναφέρετε προσθέσετε και την κατηγορία των ηλικιωμένων θα συμπληρώνατε νομίζω τον κατάλογό σας. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος στο 35. Εγώ νομίζω πως είναι δίκαιο. Εγώ προέρχομαι από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Είναι σωστό να συνεχίζουμε να τονίζουμε τα οικονομικά ζητήματα και πιο ειδικά θέλω να αναφέρω το συγκεκριμένο σημείο των εμπορικών ισοζυγίων και των μακροοικονομικών διαφορών ανάμεσα στις χώρες. Αυτό που συνέβη στην περίοδο πριν από την κρίση είναι ότι ίσω υπερβαλικά μεγάλη εμπιστοσύνη ελευθερία ε, στην, στην εμπιστοσύνη στην αγορά. Ότι δηλαδή η αγορά μπορεί μόνη να ρυθμίσει τα κακό σκήμενα του κόσμου. Και η στάση των διαφόρων κυβερνήσεων για χρόνια ήταν να παρεμβαίνουν όσο γίνεται λιγότερο, ελπίζοντας ότι λόγω της οικονομικής ανάπτυξης ε, η φτώχεια θα αρχίζει να μειώνεται. Συνέβη αυτό και υπάρχουν έχει απόδειξη ότι σε ορισμένε περιοχέ του κόσμου συνέβη όντω αυτό, αλλά στην πράξη δεν συνέβη στο βαθμό που περίμενε ο κόσμο. Γιατί σε μια κατάσταση ελεύθερης ε, αγοράς υπήρξε ε, χειραγώγηση. Τα αποτελέσματα, χωρίς να μπω τώρα σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχω χρόνο, ότι σημαντικές χώρες, η Κίνα, πιο συγκεκριμένα η Γερμανία, η Ιωπανία, οι χώρες αυτές συγκέντρωσαν τεράστια σε πλεονάσματα, τα οποία δεν συνέβησαν έτσι τυχαία, συνέβησαν, υπάρχουν γιατί υπήρξαν πολύ συγκεκριμένες παρεμβατικές πολιτικές αν αυτές οι μακροοικονομικές ε, διαφορές δεν διορθωθούν με πολύ συγκεκριμένη παρέμβαση αυτή τη φορά από τις κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων ε, περιφερειακών ρυθμίσεων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα γίνεται πλέον ε, χειραγώγηση, γιατί αν αυτές οι διαφορές δεν λυθούν με διεθνείς ρυθμίσεις, τότε η εναλλακτική λύση είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Λαμβάνουμε ένα σωρό μέτρα για να περιορίσουμε τις διαφορές και δράσεις όπως γίνονται σε διάφορες χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι λιγότερα χρήματα για την ανάπτυξη Όλα ένα και περισσότερες μεταρρυθμίσεις, αλλά ε, πρέπει να γίνουν, θα γίνουν. Πρέπει να τονίσουμε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ώστε να μην να ενεργοποιηθεί η αγορά εργασίας, περισσότερος κόσμος να έχει ευκαιρίες. Εάν δεν αρθούν οι περιορισμοί στην εσωτερική αγορά, αυτό δεν θα γίνει και έπειτα μια μεγάλη προσπάθεια για τη διόρθωση των διαφορών και να αναγκαστούν αυτοί οι οποίοι κέρδισαν ανεπίτευτα πλεονάσματα εις βάρος των άλλων χωρών να διορθώσουν την κατάσταση. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε όλες οι άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων το πιο αδύναμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα περισσότερη φορολογία, περισσότερη φτώχεια, περισσότερη ενεργεία ε, προ όφελο άλλων. Άλλοι χαίρονται ε, και υποφελούνται, ενώ οι φτωχοί συμπεριλαμβανομένων αυτών στην Ισπανία, την Πορτογαλία και άλλων στην Ευρώπη θα, ε, αυξη... θα... θα δουν να αυξάνονται οι φτωχοί τους. Ευχαριστώ κύριε στο 249. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είμαι ο Λίντο Χόρμανς, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά τις Στόχες. Είναι ένα δίκτυο εθνικών δικτύων σε κάθε κράτος μέλος και ευρωπαϊκών οργανώσεων που εργάζονται στην καταπολέμηση της φτώχειας. Έχουμε και μια συμμαχία ΜΚΙΟ. Για... Είχαμε συμμαχία για το έτος 2010 Ενδιαφέρον είναι μια που βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βοηθάμε σε αυτή την αγορά πολιτών. Να πούμε Ακούσαμε τα σχέδια της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την Ευρώπη 2020 και ειδικά την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της ε, φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αλλά αυτό το οποίο δεν υπάρχει και το είχαμε πει και νωρίτερα είναι πως τώρα που δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στα κράτη-μέλη και αναμένουμε τόσα πολλά από αυτά, βλέπουμε πως ε, αυτά τα οποία γίνονται τα μέτρα λαμβάνονται περισσότερο στο ευρωπαϊκό επίπεδο και βλέπουμε λιγότερη ανάμειξη, η πίεση, η πρόσκληση προς τα κράτη-μέλη να οργανώσουν εθνικό διάλογο για την καταπολέμηση της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω μια έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωβουλευτές και στις Επιτροπές του Κοινοβουλίου να επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για να οργανώσουν μια εθνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της φτώχειας και να οργανώσουν και εθνικές πλατφόρμες κατά της φτώχειας, στις οποίες οι φτωχοί θα έχουν ε, έναν σημαντικό ρόλο. Και βλέπουμε τώρα πως ε, υπάρχει μια συνάντηση τέτοιων ανθρώπων και θα γίνει και επί Προεδρίας και ελπίζουμε αυτό να είναι μια αρχή ώστε οι εθνικές πλατφόρμες ε, κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού να μπορέσουν να υποστηριχθούν ε, και με κονδύλια, χρηματοδότηση, ευκαιρίες ε, με το να προσκληθούν σημαντικοί ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν σε αυτές τις εθνικές πλατφόρμες έτσι ώστε όσοι έχουν εμπειρία της φτώχειας να μπορούν να λάβουν μέρος στη συζήτηση των πολιτών και αυτό να γίνει και από πραγματικούς πολίτες στο κάθε κράτος μέλος. Ελπίζω να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επηρεάσει την κατάσταση και ως προς την Κομισιόν και το Συμβουλίο. Ευχαριστούμε κύριε Χόρμαντς. Ο κύριος Σιγκουέιρα. Πολύ σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλημέρα σας. Είμαι από την Πορτογαλία. Είμαι συνδικαλιστικός ε, ηγέτης ε, και μέρο ε, της Εθνικής Επιτροπής. Βρισκόμαστε σε μια φάση που πρέπει να ξαναδούμε κάποια ιστορικά θέματα για τη φτώχεια. Η φτώχεια σήμερα παίρνει πτυχέ που είναι διαφορετικές, έχει διαφορετικά πρόσωπα και μέσω αυτού του φαινομένου επηρεάζει όλη την κοινωνία. Ακόμα και εκείνες τις κοινωνίες που θεωρούσαν και ε, προανήγγυλαν ότι είναι οι πιο ανεπτυγμένες. Σήμερα υπάρχουν πολίτες που για την θέση απασχόλη τους ε, βρίσκονται στο ε, κατόφλι της φτώχειας. Παίρνει νέε μορφές ε, η φτώχεια και τομείς της κοινωνίας που ποτέ δεν είχε φανταστεί κανείς εγγράφονται μέσα σε αυτή την έννοια της φτώχειας και βρίσκονται σήμερα ένα βήμα από το να εγγραφθούν στη φτώχεια. Το, το θέμα που θέτω είναι πολύ απλό και άμεσο. Διαρωτώ με πώς είναι δυνατόν τρία χρόνια μετά, μετά από αυτή την κρίση καμιά πολιτική εξουσία εξουσία στο παγκόσμιο επίπεδο να μην έχει προτείνει να ληφθεί κανένα μέτρο όσον αφορά την κατάργηση των φορολογικών παραδείσων. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος το 138 παρακαλώ. Ε, good morning. Ε, καλημέρα, καλημέρα σας. 138 πρώτα και μετά εσείς παρακαλώ. 138 πρώτα. Ευχαριστώ. Mm, Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ εκπροσωπώ το Φόρουμ Αλληλεγγύης ε, για την Ευρώπη Φόρουμ Αλληλεγγύης. Εκπροσωπούμε και αρκετά πολωνικά δίκτυα, καθώς επίσης και διεθνή δίκτυα. Επίσης ενδιαφερόμαστε στα θέματα που αφορούν τους μετανάστες στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Αλλά επίσης εκπροσωπούμε και ένα ίδρυμα για την αλληλοβοήθεια. Και ακούσαμε πολλές παρεμβάσει. Ε, και απόψεις να εκφράζονται. Πολλά ακούγονται και δραματικά μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι προγράμματα και σχέδια σε εθνικό επίπεδο ουσιαστικά θα έχουν αηφόρο αποτέλεσμα σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, χρονορίζοντα. Διότι φοβούμε ότι κάποια από αυτά τα σχέδια, αρκετά από αυτά τα σχέδια, ουσιαστικά δεν βοηθούν χειροπιαστά αυτούς που έχουν τόσες ανάγκες. Διασπαθίζονται πολλά κονδύλια και σε μεγάλο βαθμό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πολλές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν στόχο να βοηθήσουν χειροπιαστά εκείνους που χρειάζονται βοήθεια. Υπάρχουν πολλά σχέδια που προωθούνται και εμφανίζονται πολύ θελκτικά, ελκυστικά σε διεθνές επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο όμως απειλούνται αυτά τα σχέδια και προγράμματα. Απειλούνται επειδή υπάρχει πολύ ισχυρό, πολύ έντονο ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών τέτοιων σχεδίων ή προγραμμάτων. Και πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ξεκινήσει και να αναλάβει μια πρωτοβουλία ώστε να δημιουργηθούν προγράμματα και σχέδια για την κοινωνική ολοκλήρωση και ένταξη όσο το δυνατόν πιο γοργά. Και στο πρόγραμμα Equal επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εισαγάγει συγκεκριμένες ε, διατάξεις και προδιαγραφές σε καινοτόμα προγράμματα για να εξοικονομηθούν κονδύλια και να μην διασπαθίζονται που όπως, πολλές φορές, προανέφερα πολλές φορές ε, γίνεται πολύ κακή χρήση και διασπαθίζονται αυτά τα κονδύλια διότι πολύ συχνά δεν στοχεύουν ε, σε εκείνες τις ομάδες και εκείνους τους στόχους ε, που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και έχει τη μεγαλύτερη σημασία να βοηθηθούν. Ευχαριστώ από το δίκτυο κατά της στόχιας. Θα μιλήσω στα τσεχικά στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι πρόκειται και για ένα θέμα, το άλλο θέμα το οποίο δεν έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα σε σχέση με την κρίση Πρόκειται για το θέμα της υπερχρέωσης, το θέμα του να, είναι, να έχει κανείς χρέη. Όχι μόνο εταιρείε ε, είναι υπερχρεωμένες, αλλά και πολίτες έχουν χρέη. Η πείρα μας δείχνει στην δημοκρατία της Τσεχίας ότι πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και να προσέξουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να εκπαιδεύονται οι πολίτες για τα οικονομικά θέματα. Πρέπει να δείχνουμε στους πολίτες μας και να μαθαίνουν εκείνοι από αυτά τα διδάγματα πώς θα μπορούσαν να προστατευθούν όσον αφορά την ε, ανάληψη ε, χρεών και να μην πέσουν στην παγίδα του χρέους. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά κάθε άτομο, κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και έτσι λοιπόν αυτό το πρόβλημα φαίνεται ότι θα είναι ένα όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στο μέλλον. Ας το συζητήσουμε λοιπόν και αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Σφάτς, λέει ο πρόεδρος. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ε, Υπότιτλοι Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, Πιέρ Ζαν Κούλο, είμαι μέλο τη Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Αντιπροσωπεύω μια οργάνωση εργαζομένων τη Γαλλία και θα ήθελα να επιστήσω εντόνω την προσοχή τη ε, συνέλευση στι ε, ε, δραματικέ συνέπειε τη κρίση όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια. Είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε συχνά, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό σήμερα. Να αναφέρω μία χώρα από τι 27, Γαλλία ο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς 110.000 σπιτικά ε, είδαν να κόβεται το φυσικό αέριο. Δεν πλήρωσαν τον λογαριασμό τους για λόγους φτώχειας. Δεν, ε, σε, σε άλλα 160 νοικοκυριά κόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή 3-4 εκατομμύρια οικογένειες πέρυσι για λόγους φτώχειας στερήθηκαν είτε την ε, τον ηλεκτρισμό ή την θέρμανση. Δηλαδή μια εξωπρεπή ζωή στερήθηκαν. Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει να, καλέ, να, να καλέσει τόσο τους νομοθέτες όσο και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αλλά και τους πολιτικούς να συσπηρωθούν, να βρουν τις λύσεις για να καταπολεμήσουν αυτή τη φτώχεια, αυτή την ε, ενεργειακή ε, ε, προσωρινή κατάσταση. Γιατί όταν κανείς δεν έχει ηλεκτρικό στο σπίτι του, καταλαβαίνετε ότι όλα τα υπόλοιπα έπονται. Θέλουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα και όχι μια απάντηση κομμάτι προς κομμάτι και γειτονιά προς γειτονιά, χώρα προς χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει λύσεις, είτε δεν ξέρω, κοινωνικά, πιο κοινωνικά τα, τα τιμολόγια, είτε μια ανασπίδα, είτε κοινωνική παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Ε, αυτό έχω να σας πω εγώ ως ε, μια έκκληση αλλά και μια έκκληση για συσπήρωση όλων των εμπλεκομένων μερών για αυτή την κατάσταση που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνη. Τρία I Ονομάζομαι Σον Χίλι από μια οργάνωση που ονομάζεται Κοινωνική Δικαιοσύνη Ιρλανδίας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την ΟΚΕ γιατί εξετάζουν αυτά τα θέματα της σημερινή κρίσης και τις στόχες ε, αυτή τη στιγμή. Γιατί πιστεύω πως ε, η Ευρώπη εν γέννη βρίσκεται σε πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Και γιατί το λέω αυτό, διότι Πολλές από τις πολιτικές που επιδιώκονται για να λύσουν ή να αντιμετωπίσουν την κρίση σε πολλές διαφορετικές χώρες μας και σε κάποιες περιπτώσεις και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζουν σε τεράστιο βαθμό τους στοχούς ανθρώπους και προκαλούν επιπλέον προβλήματα σε αυτά που ήδη είχαν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα προβλήματα πιέζουν τους, τους ανέργους, τους ε, φτωχούς εργαζόμενους και για τους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα μπει στον ε, αγορά εργασίας. Είναι πολιτικές που μετακινούν πόρους μακριά από τους φτωχούς για να επιστρέψουν ε, τους πόρους αυτούς στις τράπεζες και στους ανθρώπους που είναι εξαιρετικά πλούσιοι και που ξεπερνούν επιπλέον στις κρίσεις τις διαδοχικές. Αυτό που συμβαίνει ε, λοιπόν έχω την εντύπωση πως οι πόροι μετακινούνται από τους στοχούς ανθρώπους που δεν είχαν ούτως ή άλλως ε, μερίδιο στην πρόκληση της κρίσης για να εξασφαλίσουν ότι άλλοι άνθρωποι θα βολευτούν οι οποίοι δεν πλήττονται κιόλα από την κρίση. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι δηλαδή. Και αν δεν αντιμετωπιστεί σύντομα αυτή η κατάσταση, πολύ, πολύ σύντομα πιστεύω πως θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ζημιώνεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο εξαιρετικά σοβαρά. Γιατί δεν δεν γίνεται κατανοητή η αλληλένδετη φύση της, της οικονομικής πολιτικής με την κοινωνική πολιτική και την περιβαλλοντική επίσης πολιτική. Νομίζω λοιπόν πως μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα θα χρειαζόμασταν δείκτες και θα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε δείκτες που θα μας ε, δείξουν κατά πόσο κάνουμε, σημειώνουμε πρόοδο και κυρίως να μας εξασφαλίσουν ότι δεν επιβαρύνουμε επιπλέον τους στοχούς ανθρώπου που ούτως ή άλλως δεν έχουν τους πόρους για να ανταποκριθούν και δεύτερον δεν προκάλεσαν αυτή την κρίση την οποία διανύουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία 148. Λέγομαι Μάρτο Μάτης και εκπροσωπώ το πρόγραμμα ανάπτυξη του ΟΗΕ. Είμαι Ουγγαρέζα όμω και θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να μιλήσω τη γλώσσα μου. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι το ότι πάρα πολλοί ομιλητές ανέφεραν ήδη πως έχουμε νέες μορφές φτώχειας λόγω της ε, παγκόσμιας κρίσης. Θα ήθελα να προσθέσω πως ε, όλες οι έρευνες ε, ε, τις οποίες έχω δει εγώ τα τελευταία δέκα χρόνια και στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη δείχνουν πως οι νέες μορφές φτώχειας εμφανίζονται στις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκίνησαν την εποχή της ένταξης και όχι με την κρίση. Σημαντικό λοιπόν είναι να το πούμε αυτό και να το γνωρίζουμε γιατί αυτό θα επηρεάσει την μελλοντική ε, στρατηγική. Καθώς είναι σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των ε, νέων και των παλαιών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διδαχτούμε από τα λάθη που κατέληξαν στο πλαίσιο των παλιών προγραμμάτων στο να έχει επιδεινωθεί η κατάσταση των φτωχών στις ε, νέες χώρες αντί να βελτιωθεί ειδικά στις περιοχές της υπέθρου. Το άλλο θέμα είναι το ζήτημα τον ε, Ρωμά και το πώς ζούνε. Όσοι δεν ζουνε σε κοινότητες ε, Ρωμά δεν γνωρίζουν το γεγονός πως ε, τα στερεότυπα είναι λανθασμένα. Σημαντικό θα ήταν να σκεφτούμε για την στρατηγική των Ρωμά το πώς ε, θα μπορέσει να συμπάρξει η μειονότητα με την πλειονότητα και βεβαίως αυτό συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη των κοινωνιών που ζουν ε, στη φτώχεια και όχι μία στρατηγική που θα τους κρατάει πάλι χωριστά. Ίσως με θετικό τρόπο αλλά χώρια. Το τρίτο ζήτημα είναι πως ε, το Περιφερειακό Κέντρο του Προγράμματος Ανάπτυξης ε, του ΙΕ στην Πρατισλάβα που αφορά τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προετοίμασε στα μέσα της δεκαετίας του 90 μία μελέτη, μία έρευνα για τους Ρωμά και αυτό θα επαναληφθεί και φέτος. Και συνεργαζόμαστε ήδη με συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να τους ενημερώσω πως αυτό συμβαίνει. Ελπίζω αυτή η έρευνα να συνεισφέρει να αποκτήσουμε μια σαφέστερη εικόνα για το θέμα αυτό. Το τελευταίο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι πως ε, κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής ε, Προεδρίας πολλές ε, οργανώσεις ήρθαν σε επαφή μαζί μου ζητώντας από το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ να τις βοηθήσει να βρουν οργανώσεις στις νέες χώρες, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που θέλουν να συνεργαστούν στην επεξεργασία της νέας στρατηγικής για τους Ρωμά. Οπότε, θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους οργανώσεων που θέλουν να μπουν σε αυτή την προσπάθεια να μας συναντηθούν μαζί μου στο μεσημεριανό. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ακόμη 15 ομιλητές στον κατάλογο, αλλά ο χρόνος πιέζει. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να γράψετε το όνομα στο έντυπο να μας δώσετε το έντυπο και θα λάβετε αύριο τον λόγο πρώτη. Λοιπόν, έχουμε τη Mercedes Bresso εδώ πέρα, αλλά νομίζω σημαντικό είναι οι τρεις μας εδώ πέρα να απαντήσουμε κάποιες από τις ερωτήσεις σας και από τα ζητήματα τα οποία θίξατε. Ας ξεκινήσω εγώ. Όπως βλέπουμε από τη συζήτησή μας, από την συνεισφορά, τις συνεισφορές σας, όταν μιλάμε για τη φτώχεια δεν είναι μονοδιάστατο το ζήτημα. Η φτώχεια έχει πολλές όψεις. Υπάρχει οικονομική κρίση, γιατί όπως αναφέραμε έχουμε πάνω από 23 εκατομμύρια ανέργους, 7 εκατομμύρια περισσότερους από ό,τι πριν από την κρίση και βεβαίως αυτό επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους που πέφτουν στην παγίδα της φτώχειας. Εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται με μερικό ωράριο. Αυτό επηρεάζει νέους ανθρώπους, π.χ. στην Ισπανία ή στη Λετωνία μιλάμε για ένα 40-50% των νέων που είναι άνεργοι. Αλλά αφορά και ανθρώπους μεταξύ 50 και 60 όταν χάνουν τη δουλειά τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν άλλοι. Αφορά τους ηλικιωμένους, όπως αναφέρθηκε, αφορά τις γυναίκες, τα παιδιά Έχουμε 20% των παιδιών στην Ευρώπη που μεγαλώνουν χωρίς να έχουν τα απαραίτητα κοινά εφόδια όσον αφορά π.χ. τη χρήση υπολογιστών, αλφαβητισμό κτλ. θα τους χρειαστούν όταν θα μεγαλώσουν. Επίσης, η οικονομική κρίση. Πράγματι, πολύ άδικη, αν δούμε την Ιρλανδία ω παράδειγμα. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη από πλευρά προπολογισμού. Όταν ήταν παχέ οι είχε ε, ισορροπημένο προπολογισμό. Οι Ιρλανδοί δούλευαν σκληρά, αλλά... αλλά... Αυτό το οποίο παρέβλεψαν οι Ιρλανδοί και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ήταν η επίβλεψη των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Έσκασαν οι κερδοσκοπικές φούσκες, είτε ήταν τα ακίνητα, είτε ήταν το χρηματιστήριο ή, άλλων, ή άλλες επενδύσεις. Χρεοκόπησαν οι τράπεζες και το Ιρλανδικό κράτος τη εγγυήθηκε και όλοι οι Ιρλανδοί φορολογούμενοι, σκληρά εργαζόμενοι και φτωχοί, ε, ξεπληρώνουν αυτό το χρέος. Και έρχομαι άρα στο ρόλο όχι μόνο των Ιρλανδικών ε, πολιτικών θεσμικών οργάνων αλλά επειδή ζούμε σε μια αγορά ενιαία και στο ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων γιατί είπε κάποιο πω δεν είναι σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγώ θα έλεγα το ακριβώς αντιστοιχό επειδή είμαι βουλευτή. αλλά όταν ζούμε σε μια κοινή αγορά όταν οικοδονούμε μια ενιαία Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων όταν πρέπει να ανταγωνιστούμε με τη Βόρεια Αμερική, με την Ανατολική Ασία. Πρέπει να συνεργαστούμε και επειδή στο Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων νομοθετούμε, ναι, πρέπει να έχουμε πολύ σκληρότερους κανόνες και νόμους ε, και για την επίβλεψη Πέρσι, παραδείγματος χάρη, πέρασε νομοθεσία για τη δημιουργία τριών νέων πανευρωπαϊκών εποπτικών οργάνων. Κάποιοι μπορεί να πείτε πως δεν επαρκεί. Τι θα γίνει με τη φορολογία, με τους φορολογικούς παραδείσους. Συμφωνώ πλήρως, αλλά η νόμη αυτή είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής διαδικασίας και συμβιβασμών. Και να έχουμε κάποιες χώρες, κάποιες κυβερνήσεις, θα αναφέρω τη Βρετανία, αλλά και τη δική μου, τη Τσεχία, όπου η πολιτική είναι κατά οποιασδήποτε μορφής ρύθμισης των χρηματαγορών. Οπότε η νομοθεσία που περνάει είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού. Κάποιοι από εμά θα ήθελαν πολύ σκληρότερους κανόνες και για, την ε, φορολογία, για τις φορολογικούς παραδείσους. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Θα δώσω το λόγο και στους για να απαντήσουν. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι πως είναι ένα πολύ διάστατο πρόβλημα, περιλαμβάνει πολλά τμήματα του πληθυσμού, είτε είναι οι μειονότητες, οι Ρωμά, όπως είπε η κυρία από την Ουγγαρία, σε κάποια από τα νέα κράτη-μέλη είναι ένα πρόβλημα πολύ συγκεκριμένο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένη στρατηγική. Ε, οι μετανάστες, η δεύτερη ομάδα εργασίας, ε, μετανάστες εντός της Ένωσης αλλά και εκτός της Ένωσης. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που θα συζητήσουμε στην ομάδα εργασία και θα το συζητήσουμε αύριο το πρωί. Τώρα θα δώσω τον λόγο στη συνάδελφο την Ιζαμπέλ Ντιρόντ και στον Σέπανελσιν. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη γιατί πιστεύω ότι πολλά πράγματα έχουν ήδη υποθεί και η δουλειά αυτή τη αγορά μόλι ξεκινά. Να πω αυτό που ρωτήσατε πριν από λίγο. Αν το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να παραμείνει παρατηρητή για όλα αυτά τα θέματα. Προφανώ και όχι, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε οργανώσει ε, την ε, συνεδρίαση αυτή διαπίστωσα ότι έχετε την εντύπωση ότι δεν εργαζόμαστε για τις μεγάλες πολύτεκνες οικογένειες, για τους ηλικιωμένους, τους Ρώμα και προσοχή στη διατύπωση. Δεν είναι η Ρώμα που είναι το πρόβλημα, είναι συχνά η δικιά μας ματιά στους Ρώμα. Αυτά τα τρία, αυτές τις τρεις ομάδες θα τις συζητήσουμε το απόγευμα στα διάφορα εργαστήρια και είναι πολύ σημαντικό εσείς να υποβάλλετε αιτήματα ή προτάσεις για αυτά αυτές τις ομάδες ανθρώπων. Μετά μιλήσατε για τους φορολογικούς παραδείσους, την υπερχρέωση των ανθρώπων, την ενεργειακή φτώχεια, τους δείκτες που θα έδειχναν ότι οι φτωχοί δεν, να, να μην πληρώσουν δύο φορές την κρίση ενώ δεν ευθύνονται οι ίδιοι για τα όσα συνέβησαν. Το θέμα των γεωργών, του κόσμου της υπαίθρου που είναι εξαιρετικά σημαντικό και την ενσωμάτωση των πολιτικών μεταξύ τους ώστε να γίνει κάτι πιο συνεκτικό και όχι κατακαιρματισμένο. Και αυτό που υπόθηκε για τους ε, αστέγους και χαιρετίζω τους ε, μουσικούς εδώ που είναι άνθρωποι που ακόμα ζουν ε, στο δρόμο και που για τους οποίους μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα ή τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν, θε, δεν ζουν πάντα όπως εμείς, χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις αλλά δεν είναι όλοι ευθυγραμμισμένοι στα ίδια πρότυπα. Όλα αυτά τα ερωτήματα σας προτείνω και εγώ τα έχω σημειώσει να τα στείλουμε στα διάφορα μας εργαστήρια. Τα εργαστήρια δεν ε, διοργανώνονται για να επανεφεύρουν τον τροχό. Τα σημειώσαμε όσα μας είπατε και θα πούμε στους Προέδρους να, ότι το ζητούμενο είναι να κάνουν συγκεκριμένες λειτουργικές προτάσεις που να απευθύνονται σε εμά τους Ευρωβουλευτές και που θα επιτρέψουν να υπάρξει συνέχεια ανά ε, ανά ερώτηση. Δεν μπορούμε εγώ και ο κύριος Ρούτζεκ να σας υποσχεθούμε το ρούνο ουρανό μετάστρα. Η αγορά του Ευρωκοινοβουλίου δεν πρόκειται να αύριο να εκριζώσει τη φτώχεια. Αντίθετα, μπορούμε να δεσμευτούμε για συγκεκριμένα θέματα για τα οποία μπορούμε να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε εδώ μια συνέχεια. Και στην ε, ΟΚΕ επίσης. Οπότε, να παραπέμψουμε όλα τα ερωτήματα στα διάφορα εργαστήρια για να βγουν από εκεί οι συγκεκριμένε προτάσει που θα μα δώσουν εμά μέσα και εργαλεία για να συνεχίσουμε τη δουλειά μα μετά την Παρασκευή. Σα ευχαριστώ πολύ. Σύντομα. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό το ότι τώρα μπορούμε εδώ να έχουμε μια τόσο γενική και καλή πλήρη συζήτηση για τα θέματα τα οποία θα τύχουν συνέχεια στις μικρές ομάδες εργασίας και που αύριο θα συνοψιστούν τα συμπεράσματα ενώπιόν μας είναι προσωπικά για μένα πραγματικά θα έλεγα απίστευτο ότι τα κράτη-μέλη δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να επιλύσουν τα προβλήματά τους μόνα τους. Είναι κάτι το οποίο μας κάνει να νιώθουμε ντροπή. Είναι πραγματικά έσχωστο ότι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χρονική συγκυρία είμαστε, ε, δίνουμε μια τόσο αρνητική εικόνα και δεν τα καταφέρνουμε. Και όσον αφορά τις μελλοντικές ε, εξελίξεις. Ε, υπάρχουν πολλές συζητήσεις ε, όσον αφορά το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και σε σχέση με τους προέδρους μας γνωρίζουν πολύ ακριβώς, επακριβώς τι πρέπει να γίνει. Όπως και η κυρία Ιζαμπέλ για παράδειγμα, ότι αυτό το σώμα ε, θέλει να διεξαχθεί μια σε ανοιχτά πλαίσια ευρύτερη συζήτηση. Αυτό είναι ένα καλό σημείο, ένα καλό μήνυμα και είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει κάτι το ίδιο και ακόμα και αν δεν είναι δυνατόν όλα να ενταχθούν μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διότι δεν υπάρχουν αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί παντός του επιστητού πρέπει παρόλα αυτά όλα τα θέματα να μπορέσουμε ανοιχτά να τα συζητήσουμε και κάτι να μπορέσουμε να κάνουμε στο τέλος τέλος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η τα κοινωνικά θέματα ε, σε σχέση με τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να μας κινητοποιήσουν και να ευρεθούν στο επίκεντρο. Αλλά διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να αυτή την πορεία να ακολουθήσουμε ε, και στα κράτη-μέλη μας. Κάτι πρέπει να γίνει στα κράτη-μέλη και να διαρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι στις περιφέρειές μας. Πώς μπορούμε όλα αυτά τα μηνύματα να τα περάσουμε προς τα έξω και χειροπιαστά να εφαρμοστούν. Χαίρομαι και προσβλέπω στι συζητήσει στις ομάδες εργασίας και χαίρομαι που θα συναντηθούμε αύριο πάλι. Και πάλι επαναλαμβάνω θερμές ευχαριστίες προς την χοροδία που τραγούδησε πριν. Ευχαριστώ. Μερσέντες Μπρένσο, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής των ε, Περιφερειών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την μπάλα που μου ρίξατε στο γήπεδό μου με τα τελευταία λόγια του Πρόεδρου Νίλσεν. Να ευχαριστήσω που μας καλέσατε και βλέπω στην πρόσκληση αυτή την ε, σημασία και την αναγνώριση της σημασίας ε, της περιφερειακής ε, διάστασης στην καταπολέμηση της στόχιας και ταυτόχρονα για το κρίσιμο ρόλο που μπορεί να παίξει και ήδη παίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην, στην, στον αγώνα για την κοινωνική ένταξη. Ο αγώνας αυτός περνά βεβαίως από την εγγύηση των εισοδημάτων των φτωχότερων εξημών, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε περνά επίσης και από μια καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας παιδείας, στέγασης, μεταφορών και ενέργειας. Και αυτά είναι θέματα των τοπικών αρχών. Το 2010 μας επέτρεψε να δώσουμε περισσότερη ορατότητα στα όσα συμβαίνουν επί τόπου με την ευκαιρία του φόρουμου που διοργανώσαμε ως Επιτροπή Περιφερειών τον Απρίλιο προσπαθήσαμε εκεί να συγκεντρώσουμε πολλέ ε, καλές πρακτικές με την συγκεκριμένη και άμεση στήριξη των μελών μας ώστε ο καθένας από εμά να μπορέσει να δει τι γίνεται καλύτερα σε άλλες πόλεις και περιφέρειες και άρα να βελτιώσουμε την δυνατότητα παρέμβασης για την ε, φτώχεια. Κάθε μια από τις τέσσερις πολιτικές ομάδες της ε, Επιτροπής ε, Περιφερειών έκανε το ίδιο και τα σεμινάρια που έγιναν από τα δίκτυα των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις αίθουσές μας ήταν πολλά. Ε, βεβαίως βλέπουμε ότι όλα αυτά δεν είναι παρά μια σταγόνα στο νερό σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί στις περιφερειές μας και στις πόλεις μας, ώστε οι κοινωνίες μας πραγματικά να είναι πιο ανοιχτές. Ε, ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά τη στόχη. Έτσι ολοκληρώθηκε το έτο και ένα, είναι μια από τι πρωτοβουλίε φάρου τη ε, ε, προσπάθειες αυτής. Είναι πολύ σημαντικό ε, το ότι μία εξ αυτών των πρωτοβουλειών ε, αφιερώθηκε στην φτώχεια. Η Επιτροπή Περιφερειών προετοιμάζει σχετική γνωμοδότηση για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να σας πω ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία για αυτή την πλατφόρμα. Χαιρετίζουμε θετικά την σαφή αναφορά του ρόλου ε, του ενδιάμεσου, του διαμεσολαβητή της Επιτροπής των Περιφερειών για να κινηθεί η κοινωνική αλληλεγγύη και να συνεχίσει η εταιρική σχέση κατά πολέμηση της, ε, του αποκλεισμού και επίσης ε, μιλάμε για τις περιφερειακές προσπάθειες που προωθούμε για να υλοποιηθεί η Ευρώπη 2020. Προτείναμε δηλαδή να υπογραφούν σύμφωνα περιφερειακά και εδαφικά. Επίσης θέλουμε να βασιστούμε σε κάποιες εμπειρίες για το σύμφωνο για την ε, συμπερίληψη και ε, τα εδαφικά σύμφωνα για την απασχόληση που ήδη έχουν ξεκινήσει για να γίνουν τέτοια σύμφωνα για το σύνολο των στρατηγικών της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Δημιουργεί επίσης μια πρωτοβουλίας που συγκεντρώνει διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία για προγράμματα μικρή τοπικής κλίμακας. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο γιατί το έχουμε επαναλάβει σε κάθε ευκαιρία πως η καινοτομία μπορεί να γίνει και στον ε, κοινωνικό τομέα και όχι μόνο στον τομέα το, της ε, τεχνολογίας ε, ή τις βιομηχανίες, η καινοτομία μπορεί να αφορά και την κοινωνική οικονομία και το κοινωνικό τομέα. Και ως προς αυτό έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι η Επιτροπή μας στις 10 Μαΐου θα διοργανώσει ένα φόρουμ για τον κοινωνικό πειραματισμό οι τοπικές, ε, και το ρόλο μάλλον των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται, να καταγράψουμε τις καλές πρακτικές ε, κοινωνικού πειραματισμού, να εντοπίσουμε τι δυνατότητε δυνατότητες και να σκεφτούμε μαζί τη πρακτική εφαρμογή τους. Επίσης θα μιλήσουμε για πόρους χρηματοδότησης με την πιθανή χρήση του, του, των ταμείων εγγύησεων και όχι μόνο του Κοινωνικού Ταμείου και του Progress. Και μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση η κοινωνική οικονομία και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο καινοτομίας και κοινωνικής καινοτομίας. Πέμπτο σημείο είναι ότι η προτεραιότητα που δίνεται στην πρόσβαση των τοπικών ομάδων στα διευθυντικά ταμεία και στις γενικές επιχορηγήσεις, καθώς και η απάντηση ε, στην αντιμετώπιση της τοπικής, ε, μάλλον της φτώχειας της υπαίθρου αλλά και της αστικής φτώχειας. Αυτά όλα τα θέματα μας απασχολήσουν φέτος, αλλά υπάρχουν και άλλα σημεία που θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε, όπως το πιθανό άνοιγμα ε, με, του κοινωνικού συντονισμού, με την ανοιχτή μέθοδο δηλαδή συντονισμού με τους κοινωνικούς φορείς και άλλους ε, ε, φορείς, έπειτα η εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή της πλατφόρμας ε, σε σύνδεση με τα εθνικά προγράμματα ε, μεταρρύθμισης για τα οποία μίλησα. Έπειτα, ο τρόπος με τον οποίο θα στοχευθούν τα φαινόμενα ακραία στόχιας για τα οποία μιλήσαμε, άστεγοι και Ρώμα, καθώς και οι πιο ευάλωτες ομάδες, παιδιά, μόνες γυναίκες, ηλικιωμένοι μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, η κρίση του φινοπόρου του 2008, όπως είδατε, όπως το γνωρίζετε, έχουν, έχει πάρει διάφορες μορφές που επιδεινώνουν την κατάσταση των πιο στερημένων. Και ωστόσο και από αυτή της βάσης η Επιτροπή Περιφερειών και οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές συμμετέχουν στην καταπολέμηση του αποκλεισμού. Η σώρευση προβλημάτων σε συγκεκριμένε περιφέρειες και συγκεκριμένε κοινωνικέ ομάδε είναι ένα φαινόμενο το οποίο διαπιστώνεται εδώ και 20 χρόνια. Δηλαδή το φαινόμενο της ε, πόλωσης των άκρων δεν συνδέεται μόνο με την κρίση. Ε, και μάλιστα ορισμένοι ερευνητέ έχουν αποδείξει πω είναι μία άμεση συνέπεια της οικονομία τη γνώση και το εξηγούν με δύο τρόπου. Καταρχήν η μεγάλη μάζα της απασχόλησης των θέσεων απασχόληση που υπάρχουν σήμερα είναι κακέ θέσει κακοπληρωμένε μερική απασχόληση σύντομου χρονικού διαστήματο και κυρίω για του νέου. Έπειτα η ανακατανομή της προστιθέμενης αξίας δεν συνδέεται πλέον, δεν, δεν, γίνεται, δεν πάει πια στην δημιουργία θέσεων απασχόληση ούτε στο δημόσιο προϋπο, ε, προϋπολογισμό. Περισσότερο η προστιθέμενη αξία συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα και κυρίως στον χρηματοπιστωτικό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα διαρθρωτικό. Είναι ένα πρόβλημα διαρθρωτικό. Δεν είναι μόνο επίπτωση της κρίσης. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και στα μέτρα που θα λάβουμε, που λαμβάνουμε, για να αντιμετωπίσουμε δηλαδή το θέμα της ανακατανομής των ε, εσόδων στην φάση της ε, παγκοσμιοποίησης και της υπερίσχυσης του διδογενού τομέα. Μου ζητήθηκε να κάνω μια σύντομη παρέμβαση. Όμως, με αυτή την παρέμβαση θα ήθελα οπωσδήποτε να σας, να σας επιβεβαιώσω και να σας καθησυχάσω ότι ακριβώς ε, η Επιτροπή των περιφερειών στοχεύει αυτό το μεγάλο εργοτάξιο των ε, διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να γίνει, να γίνει περαιτέρω εξέλιξη με πιο βιώσιμο τρόπο. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Ευρώπης της 2020 ε, αυτός είναι ο στόχος αλλά και πρέπει να είναι και ο στόχος των δικών μας ε, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Γιατί αν σε αυτό το επίπεδο προσπαθήσουμε να δώσουμε συγκεκριμένα τις απαντήσεις στα προβλήματα που συζητά η αγορά ε, θα είναι πιο αποτελεσματικό. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε Μερσέντες, ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, φίλοι, οι εργασίε μα για την Ολομέλεια σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια ολοκληρώθηκαν. Σα προσκαλώ στο γεύμα, όπω ήδη προανέφερα, στον πρώτο όροφο αυτού του κτηρίου. Θα ξανασυναντηθούμε στι 2.30 το απόγευμα για την εργασία στι ομάδε εργασία, workshops. Προτού αποχωρήσουμε κάποια δελτία ε, που πρέπει να συμπληρωθούν, τον Μάικλ Μακέι ο οποίος άφησε κάπου εδώ τα χαρτιά του κιόλας. Εδώ λοιπόν, βλέπετε το έχουμε. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας όρεξη. Γεια σας.